Ξέρουμε τι μας περιμένει και πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε με θάρρος την πρόκληση αυτή. Σας ευχαριστώ και ελπίζουμε στη συνεργασία σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ωνία Σκάιτεν. Σας παρακαλώ, ε, καθίστε. Να ψηφίσουμε τώρα. για την εκλογή του διαμεσολαβητή. Παρακαλώ καθίστε. Λοιπόν κύριε και κύριοι, άρχεται η ψηφοφορία, η διαδικασία της ψηφοφορίας. Παρακαλώ καθίστε. Κυρίε και κύριοι, θα κάνουμε μία δοκιμαστική ψηφοφορία όπως και χθες για να διαπιστώσουμε εάν είναι παρόντες πάνω από τους μισούς βουλευτές στην αίθουσα. Παρακαλώ καθίστε. Είχαμε ένα κατάλογο ζωγράφων χθες, θα τους αναφέρω και σας παρακαλώ να συμμετάσχετε στην ε, ε, δοκιμαστική αυτή ψηφοφορία. Είναι η ίδια διαδικασία όπως χθες. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πέρας της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 462 Λοιπόν, 71-64, ε, κανείς δεν πήρε την πλειοψηφία. Κλίν, Φανχόχ και Ρενουάρ, μάλιστα. Και Πικάσο. Ωραία. Παρακαλώ, καθίστε. Μα περιμένω τόση ώρα. Η ψηφοφορία προβλεπόταν για τις 11.30 και είναι ήδη 11.32. Όταν είμαι πρόεδρος, ε, εγώ κύριε Λάγγεν, σεβόμεθα το χρόνο. Σε λίγο θα είναι 11.35. Ε, ωραία, να περιμένω λίγο ακόμη. entsetzlich. So. Λοιπόν, αγαπητές κυρίες και κύριοι, διαπιστώσαμε μέσω της δοκιμαστικής ψηφοφορίας ότι είναι παρόντες πάνω από τους μισούς ε, βουλευτές. Ε, αυτή τη στιγμή το διαπιστώνω και οπτικός. Να σας ενημερώσω. Οι υποψηφιότητες Μπρένιγκ Μάια και Γιέγκα έχουν αποσυρθεί. Οπότε έχουμε τους εξής υποψήφιους και υποψήφιες. Ρία Όμεν Ρόιτεν, Έμιλι Ορέιλι, Τάγμα Ροντ Μπέρεντ, Φραντσέσκο Περόνι. Θα κάνουμε τώρα το δεύτερο και ενδεχομένως τρίτο γύρο της προφορίας ε, ε, τον ένα μετά τον άλλον αμέσως. Οπότε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν έρθει. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Haben alle... Ψηφίσατε όλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Πέρας της ψηφοφορίας. Λοιπόν, ψήφισαν. 640. 48 αποχές. 321 είναι η πλειοψηφία. Κανείς δεν επέτυχε αυτή την πλειοψηφία. Ωραία. Με βάση τον κανονισμό θα γίνει τώρα ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων με τις περισσότερες ψήφους. Των δύο υποψηφίων που πήραν τις περισσότερες ψήφους στις, ε, στην δεύτερη ψηφοφορία. Είναι λοιπόν οι κυρίες Όμεν Ρόιτιν και Ο Θα προετοιμάσουμε τώρα την ψηφοφορία για αυτές τις δύο υποψηφίους υποψήφιες. Περιμένετε παρακαλώ για να ε, ε, προσαρμοστεί το σύστημα. So. Ωραία. Άρχεται τώρα ο τρίτος γύρος της ψηφοφορίας. Παρακαλώ ψηφίστε σε αυτόν τον τρίτο γύρο. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Υπάρχει κάποιος που δεν μπόρεσε ακόμη να ψηφίσει. Όχι, ωραία, πέρα της ψηφοφοριες Εψήφισαν. 635, 36 αποχές, ε, συγγνώμη, 63 αποχές, εξελέγει με 359 ψήφους η κυρία Έμιλι Ο'Ράιλι. Κυρίες και κύριοι, άρα με βάση το αποτέλεσμα της τρίτης ψηφοφορίας η κυρία Έμιλι Ορέιλι εκλέγεται Ευρωπαίος διαμεσολαβητής, της συγχαίρω και με βάση το άρθρο 204 παράγραφος 7 του εσωτερικού κανονισμού την καλό να ε, ορκιστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η εντολή της θα αρχίσει την 1η Οκτωβρίου 2013 εφόσον προηγουμένως ε, λάβει χώρα η ορκομοσία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το λόγο έχει ζητήσει τώρα ο Επίτροπος κύριος ε, Σεύκοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ θερμότατα την κυρία Οράιλη για την εκλογή της στην θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Είναι πάνω στο θεωρείο, αντιλαμβάνουμε. Συγχαρητήρια λοιπόν. Και Και φυσικά κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω το γεγονό ότι για πρώτη φορά μια γυναίκα καταλαμβάνει αυτή τη θέση του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τίτλος. Θα είναι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Αλλά η κυρία Οράιλη το γνωρίζει πολύ καλά, διότι ήταν ε, η πρώτη γυναίκα συνήγορος του πολίτη στην Ιρλανδία από το 2003. Κυρία Οράιλη, θα ασκήσετε ε, ένα πολύ δύσκολο έργο και η Επιτροπή θα είναι δίπλα σας, εταίρος σας, γιατί η Επιτροπή είναι μόνος, το μόνο όργανο που υιοθετεί τις αποφάσεις προς τους πολίτες και η Κομισιόν θα κάνει κάθε προσπάθεια να βρει ε, θετική έκβαση στις, στα προβλήματα και συστάσεις. Είναι σημαντικό μαζί να μεταφέρουμε το μήνυμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα όργανα τις, ε, ασχολούνται με τα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουν. Είναι σημαντικό οι πολίτες της Ευρώπης να αντιληφθούν ποια είναι τα δικαιώματά τους, όπως και το δικαίωμα καταγγελίας στον διαμεσολαβητή. Είναι αυτό που σημαίνει η Ευρώπη των πολιτών. Σας εύχομαι όλα τα καλύτερα για το έργο που θα αναλάβετε και θα βρισκόμαστε πάντα στο πελευρό σα με τις εξαιρετικές σχέσεις τις οποίες ήδη υπήρχαν ανάμεσα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και την Επιτροπή στο παρελθόν. Συγχαρητήρια και προσβλέπω στην μελλοντική συνεργασία μας στο μέλλον, κυρία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες για το ψήφισμα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κυρίες και κύριοι, να ψηφίσουμε πρώτα για το ψήφισμα της ομάδας των Πρασίνων. Για την παράγραφο 1 έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 63 η τροπολογία 1 έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το ψήφισμα συνολικά. Ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται το ψήφισμα. Περνάμε τώρα στο κοινό ψήφισμα ΕΛΚ, Σοσιαλιστών και ΑΛΔΕ. Μετά την παράγραφο 1, τροπολογία 15, ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 2. Τροπολογία 2. Ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ονομαστική. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 3. Τροπολογία 18. Ονομαστική. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η παράγραφος 4 του αρχικού κειμένου κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 20, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 4, ονομαστική, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Μετά την παράγραφο 6. Στην παράγραφο 6. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 ονομαστική άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται η αρχική παράγραφος 6 ονομαστική άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 6, τροπολογία 13, ονομαστική. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 14. Ονομαστική. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 24. Ονομαστική. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 25. Αναθεωρημένη. Ονομαστική. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 7 τροπολογία 6 ονομαστική άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται Τροπολογία 7. Ονομαστική. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Ονομαστική. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Νέα ονομαστική. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 12. Τροπολογία 10. Ονομαστική. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Στην αρχική παραγραφό 12 ο κύριος Κάλφιν θέλει να κάνει μια προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ. Θα έλεγα στην παραγράφο 12 να κάνουμε μια μικρή τροπολογία, δηλαδή να διευκρινίσουμε χωρίς να αλλάξουμε το νόημα της φράσης που λέει καλωσορίζει το γεγονός ότι έχει ληφθεί διατάξη για αύξηση στο ένα δις από το σχέδιο ε, το, της των τροφίμων από εκείνα τα κάτι μέλη που επιθυμούν να αλλάξουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την αύξηση αυτή την αύξηση να, προσθεθεί, να προσθεθούν αυτές οι δύο λέξεις. This increase. Θα πρέπει ε, τυπικά να ρωτήσω εάν είναι κανείς κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας. Έχει αντίρρηση να υποβληθεί. Όχι. Ωραία. Τότε να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο όπως το τροποποίησε ο συνάδελφος Κάλφιν. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στροπολογία 11. Ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η το αρχικό κείμενο της παραγράφου 13. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 13 τοπολογία 12 ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απόλυτε. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απόριπτε. Ψηφίζουμε τώρα συνολικά το κείμενο ψηφίσματος. Εάν εγκριθεί, ε, καταπίπτουν όλες οι άλλες υποβληθήσεις, ε, όλα τα άλλα υποβληθέντα ψηφίσματα. Το τροποποιηθέν ε, ψήφισμα ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται το κοινό ψήφισμα. Τώρα περνάμε στην έκθεση Μορέιρα. Την πρώτη από τις δύο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική. Πέρας. Ωραία, ωραία. Παραμένει ανοιχτή η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη δεύτερη έκθεση Μορέιρα, ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Σόουζα. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ονομαστική ψηφοφορία. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα θα πρέπει να διακοπεί η ψηφοφορία για την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ. Παρακαλώ να μείνετε στην αίθουσα.